Οπότε εγκρίνονται τα πρακτικά. Έλαβα τις θέσεις του Συμβουλίου όσον αφορά τον κανονισμό αμοιβαία στήριξη μεταξύ διοικητικών αρχών των κρατών μελών. Τον κανονισμό για το καθεστώς του δικαστηρίου, για το καταστατικό του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι τίτλοι θα συμπεριληφθούν στα πρακτικά αυτής της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η προθεσμία των τριών μηνών αρχίζει να μετράει από αύριο 10 Ιουλίου του 2015. Πρώτο σημείο στην απογευματινή ημερήσια διάταξη.